και μετά βεβαίως ένα διάλειμμα και το απόγευμα και συνέχεια το βράδυ. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευτεί σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εύχομαι καλό δρόμο και καλό ύπνο.